οτροπία στους πολίτες της χώρας, αλλά και να βελτιώσουν την κατάσταση για τους ομοφιλόφιλους, λεσβείες, διεμφυλικούς και επιφιλόφιλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Έξι προτάσεις ψηφίσματος έχουν κατατεθεί και θα γίνει η ψηφοφορία στο τέλος της συζητήσεως. Και τώρα έχουμε τους πρόσφυγες από την Ερυθρέα που κρατούνται όμοιροι στην Χερσόνησο του Παρακαλώ την κυρία Σουάλκη να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, περίπου 150 πρόσφυγες από την Ερυθρέα κρατούνται από ό,τι φαίνεται πρόσφυγες στο Σινά, στο και περιμένουν να πληρωθεί να πληρωθούν λίτρα στους λαθρεμπόρους ανθρωπίνων όντων που τους έχουν στα χέρια τους. Από το 2007 συνεχίζεται αυτό το λαθρεμπόριο στην έρημνο του Σινά. Γίνονται προσπάθειες από τις ε, αρχές του ΟΗΕ να ερευνηθούν αυτές οι καταγγελίες. Πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες της Αιγύπτου μαζί με την υπάτη αρμοστία για τους πρόσφυγες για να, καταληθούν, να καταληθούν τα δίκτυα των λαθρεμπόρων και να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο σεβασμό των διεθνών προτύπων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπερβολική βία εναντίον των προσφύγων και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε και εμείς να το τονίσουμε και για αυτά που γίνονται στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Ασάκη. Ο κύριος Σάσολη για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση στο ΣΥΝΑ. Θεωρούμε αυτά τα γεγονότα τα, για τα οποία έχουν ενδιαφερθεί ακόμα και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Κοινοβούλιο μα. Εγώ θέλω να προσκαλέσω την Επιτροπή να δείξει ενδιαφέρον ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικά κατεπίγουσα κατάσταση σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πράξουν όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν του πρόσφυγε αυτού οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από το έδαφο τη χώρα του. Εμεί θεωρούμε ότι μπορούν να τύχουν ασύλου σε ευρωπαϊκέ χώρε. Ζητάμε λοιπόν από την Κομισιόν να πράξει όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να λάβει χώρα αυτή η, η ενέργεια, χρησιμοποιώντα και τα κονδύλια τα οποία δίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο τη Πρόσφυγη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σάσολη, ακολουθεί για ένα λεπτό κύριο Στάνο. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, οι συντηρητικοί μεταρρυθμιστέ καταδικάζουν αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά ει βάρο αυτών των ε, αυτό είναι σαν να έχουμε την σημερινή μέρα ε, δουλεία. Τι έγινε. Έρευνες κάνει η κυβέρνηση όσον αφορά αυτούς τους ισχυρισμού για την απελευθέρωση των προσφύγων όμως. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους καημένους. Γιατί ε, γίνονται πρόσφυγες. Είναι διότι το καθεστώς της χώρας τους είναι από τα πιο σκληρά δικτατορικά καθεστώτα και οπότε προσπαθούν να φτιάξουν ζωή τους κάπως κάπου αλλού. Στην Ερυθρέα θα πρέπει ή να πάνε στο στρατό ή να μπορούσαν να ζήσουν μέσα σε μια οικονομία διαλυμένη από τόσους ε, πολέμους μέσα στη διαφθορά. Η Ερυθρέα δεν έχει κάνει ποτέ κοινοβουλευτικές εκλογές. Και από το Wikileaks τι, τι προέκυψε ότι υπήρχε διαπλοκή μεταξύ ξένων ε, διπλωματών και ηγετών της χώρας. Θα πρέπει να καταδικάσουμε τον τύρανο, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για ακόμα και να αναστείλουμε όλα τα προνόμια από τη Συμφωνία Κοτονού για τη χώρα εκείνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Τένο. Πρέντα είναι ο επόμενος. Κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο έχουμε χιλιάδες οι οποίοι επειδή είναι τόσο άσχημη κατάσταση στο κύριε Αφρικής φεύγουν πέφτοντας στα χέρια των δουλεμπόρων. Δεν υπάρχει κανείς σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έτσι. Βλέπουν δολάρια, βλέπουν λεφτά αντί να βλέπουν ανθρώπους αυτοί οι έμποροι. Πάμε σε κάτι τιμές περί τα 8.000 δολάρια ανά όμηρο. όπως θεωρούνται αυτοί οι άνθρωποι και έχουμε επίσης ε, τις γυναίκες που είναι ακόμα θύματα βιασμών και θα πρέπει επομένω να καταδικάσουμε αυτές τις ε, συμπεριφορές, αυτές τις ενέργειες. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η Αίγυπτος κάνει ε, προσπάθειες απελευθέρωση ομήρων και επίσης να καταπολεμήσει αυτούς τους δουλεμπόρους. Λοιπόν, ένα κράτο μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Για δύο λεπτά τώρα ο κύριο Ταβάρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση των προσφύγων στην ε, Ερυθρέα που βρίσκονται στην έρημνο του Σινά είναι πάρα πολύ σοβαρή, όπω περιγράφηκε από πάρα πολλού συναδέλφου. Προφανώ είναι απαραίτητο να είμαστε στεναροί για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε του λαθρέμπου ανθρωπίνων όντων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δει πώ λειτουργεί αυτή η διαδικασία λαθρεμπορίου. Πρέπει όμως να προστατεύσουμε και τους ε, πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε χειρώσεις στους λαθρεμπόρους και να ξεχάσουμε τα βάσανα αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει να σκεφτούμε και ποιες, ποια είναι τα αίτια που έχουν οδηγήσει τον κόσμο αυτό να περνά από το σειρά. Γιατί η οδό μετανάστευσή του προπαρελθόν ήταν μέσα από τη Λιβύη και με τι πρόσφατε συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λιβύη έχουν επιλέξει να πηγαίνουν από το Σινά. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην ε, Λιβύη είναι ουσιαστικά κέντρα στατόπεδα συγκεντρώσεως. Είναι αυτό το οποίο ονομάζεται ως η Βόρεια Κορέα της Αφρικής το έδαφος της Λιβύης. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν η οποία είναι εν μέρει υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει το ταχύτερο δυνατό μια αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο για να μπορέσει να διαπιστώσει επί τόπου ποια είναι η κατάσταση. Και εμπλέκονται όλα τα θεσμικά μα όργανα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια πραγματική πολιτική για την επανεγκατάσταση των προσφύγων αυτών. Δεν μπορούν να μείνουν στη χώρα του, δεν μπορούν να μείνουν σε μια χώρα διαμετακόμιση. Θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο να εγκατασταθούν σε χώρε αυτέ. Δεν προχωράει το θέμα αυτό όμως της επανεγκατάστασής τους γιατί το Συμβούλιο εξακολουθεί να χρονοτριβεί και να μην αποδέχεται τη χρήση του, του πακέτου για την επανεγκατάσταση και την χρηματοδότησή του. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά αυτό το πακέτο και για το θέμα αυτό είμαι εγώ ο ίδιος εισηγητής θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει ένα κατεπήγον σχέδιο για να αντιμετωπίσει το θέμα επανεγκατάσταση. Αλλά αν δεν το κάνει και το Συμβούλιο το δικό του κομμάτι στα πλαίσια τη συναπόφαση, θα παραμείνουν αυτοί στο ΣΥΝΑ για πάρα πολύ καιρό. Και αυτό σημαίνει ότι παίζονται ανθρώπινε ζωέ. Είναι καιρό στο Συμβούλιο να προχωρήσει και να κάνει κάτι για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταβάρε. 1,5 λεπτό κυρία Λόχτφιλτ. Σας ευχαριστώ. Ένα τηλεφώνημα μεταξύ ενός, ενός ιερέα Ερυθρέου στην Ιταλία και, άλλο, και ενός Ερυθρέου στην ε, Αίγυπτο ήταν αρκετό για να μάθει όλος ο κόσμος ότι κινδυνεύουν από ε, εκτέλεση οι Ερυθρέοι αυτοί οι σκλάβοι ε, εφόσον δεν πληρώσουν τα λίτρα που απαιτούν οι σωματέμποροι. Πρόκειται για απάνθρωπα εγκλήματα τα οποία διεξάγονται στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, στα οποία καταφεύγουν πρόσφυγες αναζητώντας διέξοδο προς το Ισραήλ ή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Και εάν περάσουν τα σύνορα του Ισραήλ κινδυνεύουν από στρατοδικείο. Τουλάχιστον 85 άοπλοι πρόσφυγες έπεσαν θύματα ε, πυροβολισμών και έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν τα σύνορα τους ε, πυροβόλησαν οι συνοριοφρουροί του Ισραήλ. Έχει αρχίσει τώρα το Ισραήλ να ενισχύει την φύλαξη και την επιτήρηση των συνόρων και έχει οργανώσει ένα μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων. Απευθύνουμε έκκληση λοιπόν και στις δύο κυβερνήσεις να συνεργαστούν με τα ε, με την οργάνωση για τους ε, πρόσφυγες των ΗΠΑ για να βοηθήσουν την κατάσταση αυτή. Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία το, την, στις νέες συνθήκες στις οποίες ζουν αυτοί οι πρόσφυγες οι οποίοι δεν μπορούν ούτε καν να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Πίλερ. Εκ μέρους των, ομάδων, των πολιτικών ομάδων τώρα παρακαλώ, ο κύριο Φκάτσιμαρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση αυτή με τους πρόσφυγες είναι κάτι το τρομερό. Οι αρχές της Αιγύπτου προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτή τη μάστιγα των δουλεμπόρων. Χρειάζεται να βοηθήσουμε και το Ισραήλ και την Αίγυπτο σε σχέση με αυτό το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων. Θα πρέπει να χτυπήσουν το κακό στη ρίζα του, να βελτιωθεί η κατάσταση στο κέρα της Αφρικής και στην Ερυθρέα συγκεκριμένα και στις άλλες χώρες όμως. Και έτσι να σταματήσει αυτή η υπόθεση. Αλλιώς θα υπάρχουν αυτές οι συνέπειες. Παρακαλώ, εγκρίνατε το ψήφισμα του ΕΛΚ που είναι καλύτερο από το κοινό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Θα Ακολουθεί η κυρία Γκόμης για ένα λεπτό. <clears throat> κύριε Πρόεδρο, η Αίγυπτος όχι μονάχα κλείνει τα μάτια στην τύχη αυτών των ανθρώπων για την εκμετάλλευση και τα βασανιστήρια που υφίστανται οι πρόσφυγες αυτής, αυτοί οι Αφρικανοί από τη Σομαλία και την ε, Ερυθρέα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις χώρες τους για να περάσουν στο Ισραήλ μέσω από το Σινά η Αίγυπτος τους στέλνει πίσω παρά το γεγονός ότι έχουν όλους τους λόγους να θεωρηθούν πρόσφυγες εφόσον έρχονται από χώρες όπου σοβούν τρομερές συγκρούσεις αιματήρες στην περίπτωση της Σομαλίας και στην περίπτωση της Ερυθρέας που είναι μία από τις πιο κατασταλτικές και πιο καταπιεστικές χώρες του κόσμου. Οι, οι αρχές εκεί στο Σινά και οι Ισραηλινές αρχές ασκούν μια δράση η οποία βασίζεται στο ότι πυροβολούμε ότι κινείται όταν βλέπουν τους πρόσφυγες. Αυτό είναι κατά των υποχρεώσεων που έχουν σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιμετώπιση των προσφύγων. Θέλουμε να ζητήσουμε επίση και από τι ευρωπαϊκέ αρχέ να υποστηρίξουν τη δράση τη υπο... υπάτη αρμοστία για του πρόσφυγε και υποστηρίζω αυτό που λέει ο κύριο Σταβάζ για το πακέτο για την επανεγκατάσταση των προσφύγων. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκόμε. Ο κύριος Ρινάλντι δεν έχει δείξει μύτη. Η κυρία Σαρτζεντίνη για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό. Αυτό είναι κάτι σαν ένα ράπισμα, διότι είχε προηγηθεί το προηγούμενο κείμενο. Είναι η κατάσταση πάρα πολύ σοβαρή και βλέπουμε τώρα τους πρόσφυγες από την Ερυθρέα τους οποίους τους εχμαλώτησαν και τους κρατάνε όμοιρους στο Σινά. Το ίδιο έγινε και με την Ιταλία και την Λιβύη. Είχαμε κάποιου... Έτσι γίνεται κάθε φορά με τους πολιτικούς πρόσφυγες οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν, να τρέξουν. Ε, τα πράγματα πάνε δηλαδή από το κακό στο χειρότερο. Από, πέφτουν και πέφτουν στο στόμα του λίγο αντί να γλιτώσουν. Επομένως θα πρέπει να προσέξουμε ε, όλη η οικογένεια κινδυνεύει αυτών των προσώπων. Οπότε θα πρέπει κάτι να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι και θα πρέπει να ανοίξουμε τις πρεσβείες μας κοντά στην Ερυθρέα και θα πρέπει να παράσχουμε άσυλο σε τέτοια πρόσωπα. θα πρέπει να αναγνωριστεί το ότι κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς να αναγνωρίσουμε ότι δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Τους αφήνουμε απ' έξω, τους εκθέτουμε και έτσι κινδυνεύουν. Ευχαριστώ κυρία Σαρχεντίνη και ο κύριος Πάσκα τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα σύνορα του Σινά προς το Ισραήλ έχουν γίνει ένα ε, στόπος διαφυγής των Σομαλών και Ερυθρέων σε αναζήτηση καλύτερων συνθήκων ζωής. Πέφτουν όμως θύματα των σωματεμπόρων, στους οποίους καταβάλουν διάφορα ποσά προκειμένου να τους βοηθήσουν, εξασφαλίζοντας τους ε, τα σχετικά έγγραφα να περάσουν τα σύνορα. Δεν έχουν όμως κανένα δικαίωμα εναντί αυτών των σωματεμπόρων και των συμμοριών τους. Τους αφήνουν, τους εγκαταλείπουν στη μοίρα τους, και πέφτουν θύματα αυτών που έχουν ε, πληρωθεί για να τους προστατέψουν υποτίθεται. Πρόσφατα είδαμε η διεισόμαση πόσο έχει οξυνθεί η κατάσταση. Είναι η ώρα πια με τις εμπλεκόμενες ε, χώρες να βρούμε μια ουσιαστική λύση στην κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πασκά. Κυρία Μακοβέη, παρακαλώ για ένα λεπτό. Το Δεκέμβριο, στις 7 Δεκεμβρίου, η Πατιαρμοσία των Εθνών για Πρόσφυγες εξέφρασε τις ανησυχίες της ε, για το γεγονός ότι κρατούνται όμοιροι 850 Ερυθρέοι από σωματεμπόρους ε, στο Σινά. Ε, κατανοούμε βεβαίως ότι προσπαθούν να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής, όμως κρατούνται μέσα σε κοντέινερ στις... Ε, στην έρημο και πολλές φορές υφίστανται ξυλοδαρμό αυτοί οι Ερυθρέη. Από την άλλη πλευρά το Ισραήλ δεν δέχεται να τους ανοίξει τα σύνορα. Παρακαλούμε λοιπόν το Ισραήλ να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα, να θέσει ένα τέρμα σε αυτό το σωματεμπόριο και να τους βοηθήσει να βρουν μια ε, αξιοπρεπή ε, ζωή με βάση και τις προδιαγραφές και τις αρχές του της των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Τώρα διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑ. Η κυρία Μπροσίσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα καταρχάς να σημειώσω ότι το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι αυτό το οποίο εγώ υποστηρίζω. Δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε με τις άλλες πολιτικές ομάδες ώστε να υιοθετηθεί ένα κοινό ψήφισμα και θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση στο στην Αφρική, στο στα αφρικανικά αυτά κράτη, διότι έχει διαρκώς, οξύνεται διαρκώς η κατάσταση όπως προς τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες που φεύγουν από τις χώρες τους και τώρα πέφτουν δυστυχώς θύματα από ό,τι μαθαίνουμε 850 συγκεκριμένοι των σωματεμπόρων ε, οι οποίοι τους μεταχειρίζονται και τους κρατούν όμοιρους. Είναι προφανές ότι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα λίτρα οικογένειες για να απελευθερωθούν αυτοί οι όμοιροι. Πρέπει λοιπόν να υψώσουμε τη φωνή μας και το παράστημά μας ε, και το ανάστημά μας και να δράσουμε κατά αυτών των σωματεμπόρων. Πρέπει να δεθεί ένα τέρμα σε αυτά τα σανιστήρια και να προσαρθούν στη δικαιοσύνη οι πέτοιοι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πασέσκου. Ο κύριος Σέκετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι απόλυτα σαφές και προφανές ότι εγώ καταδικάζω την κατάσταση στο ΣΥΝΑ και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για να τους προστατεύσει και να βελτιώσει την κατάσταση διαβίωσής τους. Αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνση η οποία αναφέρεται από αυτό το ψήφισμα για μένα οδηγεί σε ένα αδιέξοδο. Εγώ θεωρώ ότι είναι λανθασμένο το να δημιουργήσουμε ένα ταμείο για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες δεν μπορώ να δεχτώ όμως να παροτρύνουμε ε, περαιτέρω πρόσφυγες να έρθουν στις χώρες μας. Ήδη στην Ουγγαρία έχουμε πάρα πολλούς πρόσφυγες που δεν μπορεί να τους απορροφήσει η χώρα μου και δεν αφορά μονάχα την Ουγγαρία, αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει καταρχήν να βοηθήσουμε τους δικούς μας πολίτες, τους δικούς μας φτωχούς που στην Ουγγαρία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Και θα πρέπει να κατανοήσετε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη στομώσει από τους πρόσφυγες. Μπορούμε να διευκολύνουμε τη μετακίνησή τους, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε πια χώρες υποδοχής. Άλλους δύο θα επιτρέψουν να λάβουν το λόγο. Η κυρία Κρετού και ο κύριος Σιωπού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Περισσότεροι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί οι άνθρωποι φύγανε από ένα καθεστώ. Ε, ήταν το καθεστώ αυτό τόσο καταπιστικό και επομένω θα πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτού και το ακριβώ το, το, πιο ενισχυτικό είναι το ότι πόσο απάνθρωποι είναι η συμπεριφορά αυτών των εμπόρων και τους, ε, ε, να μην θεωρούμε ότι έτσι το πρόβλημα θα λυθεί με το να κλείσουμε τα μάτια θα πρέπει κάτι να κάνει η διεθνή κοινότητα γιατί αυτό το εμπόριο ανθρώπων, ε, των ανθρώπων από την Αφρική ε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο προσπαθούν να λύσουν οι Αιγυπτικές αρχές τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει επομένω η λαθρομετανάστευση να αντιμετωπιστεί αλλά με, διαφορετικά μέσα, διαφορετικό τρόπο. Και θα πρέπει η, η ΚΝΟΥΡ ε, ε, κάτι να κάνει ώστε να βοηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ κύριε Κρετού. Τελευταίος, κ. Τσιόρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι πρόσφυγες της Ερυθρέας αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα τραγική κατάσταση. Ενώ εμείς παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να κατανοήσουμε και γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταστολή και η καταδίωξη των πολιτικών αντιφρονούντων στην Ερυθρέα συνεχίζεται. Αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες του κακού, οι ρίζες του προβλήματος. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αλλάξουμε τη στάση που κρατάμε έναντι της κυβέρνησης της Ερυθρέας. Το 2007 ο τωρινός ηγέτης της Ερυθρέας και ο οποίος ήταν ο υπεύθυνο για την ε, αποτρόπια κατάσταση της χώρας έγινε δεκτός μεταβαίων και κλάδων στις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την αντιμετώπιση της Ερυθρέας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζιόμπρο. Για το τέλος της συζήτησης δίνω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Πίμπαλξ. Αγαπητοί κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τον προβληματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και έχουμε αυτήν την εκθεσία που μιλάει για τι εκατοντάδε των ε, ε, προσφύγων από Σομαλία, Σουδάν, Ερυθρέα που κρατούνται όμοιροι στην έρημο του Σινά και απίτησαν χρήματα για να τους απελευθερώσουν. Παρακολουθούμε αξιολογούμε και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση. Έχουμε την αντιπροσωπή μας στο Κάιρο. Έχουμε στενή συνεργασία με τις, τους τοπικούς φορείς αλλά και με την, ε, με, με την UNCHR. Υπάρχει συντονισμός και με τις πρεσβείες των κρατών μελών και Ήρθαμε σε επαφή και με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διατυπώσαμε την ανησυχία μας και το ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει η Αίγυπτος να αναλάβει δράση, να περιθερώσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους προστατεύσει όπως πρέπει. Μαθαίνουμε ότι γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν και ελπίζουμε ότι θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση μέσα μέρες. Όμως ε, δεν είναι αυτή η περίπτωση η μόνη. Γιατί υπάρχουν πολλά κενά στην προστασία των προσφύγων στη χώρα και ε, στο ΣΥΝΑ έχουν αναφερθεί πολλά τέτοια σχετικά περιστατικά. Όσοι προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα ε, υφίστανται επιθέσεις, παρενοχλήσεις και το Ισραήλ και η Αίγυπτος προσπαθούν να συνεργαστούν πάνω σε αυτό ε, και να ρυθμιστεί το θέμα και από, από, από πλευρά μετανάστευση και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει αυτή η Επιτροπή συνεργασία. Στι 14 Δεκεμβρίου έγινε μια τέτοια συνάντηση στο Κάιρο και προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή με τι αρχέ για να βελτιωθεί το σύστημα και να προστατευτούν όλοι αυτοί οι τούντε άσυλο και πρόσφυγε. Τεχνική και οικονομική αλλαγή έχει προσφερθεί. Επίση η Ένωση κάλεσε τις αρχές της Αιγύπτου να εξασφαλίσουν το ότι δεν θα επαναπροωθούνται όλοι αυτοί οι μετανάστες. Και αυτοί που έρχονται από την Ερυθρέα. Η... Ο Ήπατος ε, είπατε εκπρόσωπος επίσης ε, έχει ασχοληθεί για όλα αυτά που γίνονται στη σχέση του Σινά. Ελπίζουμε θα έχουμε κάποια, κάποιες θετικές εξελίξεις και ήδη η Αίγυπτος έχει καθυρώσει ως ποινικό αδίκημα την εμπορία ανθρώπων και έχουν θεσπιστημένες και αντίστοιχες κυρώσεις. ποινικοποίηση επίσης αφορά και το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Ελπίζουμε ότι θα ληφθούν επομένως και τώρα αποτελεσματικά μέτρα ούτω ώστε να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία. Και θα υπάρξει όσο γίνεται καλύτερη συνεργασία. Εμείς θα συνεχίσουμε να προωθούμε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ε, του, τον, τον ΟΗΕ και έτσι να η κατάσταση στη χώρα. Όσον αφορά δε τους ομήρους του, του ΣΥΝΑ θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το τι θα γίνει, θα συνεργαστούμε με τις Αιγυπτικές Αρχές και ειλικρινά ελπίζουμε τον μέτρο δυνατόν να ανεβρεθεί μια λύση και είναι πάρα πολύ θυμερό το ότι χάθηκαν οκτώ ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Πίμπαλξ. Κύριε Ταβάρης, για ένα διαδικαστικό παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μας ανέγνωσε μια ήδη έτοιμη απάντηση Επιτροπής Επιτροπή, σαν να μην έθιξε κανείς κάτι το ιδιαίτερο. Ο πρόεδρος, σας παρακαλώ να τοποθετηθείτε επί του κανονισμού, κύριε συνάδελφε. Ζητήσατε το λόγο επί του κανονισμού, να τοποθετηθείτε επί του κανονισμού και για τίποτε άλλο. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Σταβάζ. Μα είναι διαδικαστικό σημείο αυτό. Ζητήσαμε από την Κομισιόν ιδιαίτερα να δώσει μια απάντηση να μας πει αν θα στείλει μια αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και τουλάχιστον η Κομισιόν θα μπορούσε να ζητήσει να κλείσει η διαδικασία της. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφοι. Δυστυχώς δεν ήταν διαδικαστική η παρέμβασή σας. Δεν έχετε το δικαίωμα να ρωτήσετε την Κομισιόν μέσα στην κανονική διαδικασία. Έχουμε έξι ψηφίσματα τα οποία ψηφίζονται τώρα. Το τα χθεσινά πρακτικά και τα κείμενα